Chers collègues, je vous invite à gagner vos places. J'ouvre la réunion de la commission des Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Αρχίζει η συνεδρίαση τη ομάδα προπολογισμών. Ζητούμε συγγνώμη. Ζητούμε στο πρώτο πληθυντικό, πρόεδρο και συντονιστέ. Οι συντονιστέ ε, στη σύσκεψή του χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε προβλέψει, αλλά ε, ήταν μάλλον λάθος του πρόεδρου της προηγούμενης συνεδρίασης. Το σημείο 6 που ήταν να ψηφίσουμε σήμερα θα αναβληθεί για αύριο, για τις 11 παρατέταρτο. Διότι η κυρία Νεριάντα, η συγγήτρια, θα έρθει αύριο. Το σημείο 13, η κυρία Τρίπελ ε, μας είπε ότι δεν μπορεί να έρθει, πρέπει να παραμείνει σε μια άλλη επιτροπή και αναβάλλεται για αύριο το μεσημέρι. Ε, στο τέλος πρωινή συνεδρίασης και το σημείο 15 για την ε, κοινωνική Ευρώπη πρόκειται για μια πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού το 2016. Ε, αυτές είναι οι αλλαγές που προτείνω για το σχέδιο μερίσσας διάταξης. Θα ήθελα για τις 16 και 17 Μαρτίου με βεβαιώσετε ότι έχετε λάβει τα πρακτικά και ότι δεν έχετε παρατηρήσεις. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Ολοκληρώθηκε μόλις η σύσκεψη των συντονιστών και λήφθησαν οι εξής αποφάσεις. Πρώτον, θα ε, κάνει γνωμοδότηση η Επιτροπή μας για την ε, συμφωνία αλίας με τις νήσους Κουκ. Οι πράσινοι θα ορίσουν οι συγητή. Γνωμοδότηση επίσης για την έκθεση Ρέτζι για το Ταμείο Λεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αξιολόγηση, το ΕΛΚ. Θα διορίσει το που θα είναι και μόνιμος συγητής εν προκειμένου για την έκθεση ΛΥΜΠΕ για, για ένα νέο σύστημα Ισρών Εκρών. Το να λαμβάνει αυτή την έκθεση. Η κυρία Χολμάγερ ε, θα είναι η συγκήτρια. Για την αντιπροσωπεία για την Ελλάδα συμφώνησαν οι ομάδες να κοινοποιήσουμε τα μέλη που θα μετάσχουν στο κλιμάκιο μέχρι τις 10 Μαΐου. Για τις δύο αντιπροσωπείες, Ελλάδα και Λίβανος και Ιορδανία, τονίσαμε πως ε, το βασικό αντικείμενο της αποστολής ε, θα ε, αφορά στον προϋπολογισμό για να προσμετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της ε, εισφοράς από πλευράς ε, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτές τις χώρες σε σχέση με τα προβλήματα που σχετίζουν με υποδοχή, υποδοχή των προσφύγων. Ε, τώρα, για τα, τη δημοσιονομική πτυχή του προσφυγικού και της μεταναστευτικής κρίσης, Ε, τροποποιεί τη στάση μας και ε, προσδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στα στοιχεία που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό. Πράξη κατά εξουσιοδότηση επίσης για επέκταση στη Λευκορωσία των εγγυήσεων για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Προτού εκδώσουμε γνωμοδότηση, θέλουμε να ζητήσουμε δίμηνη παράταση, ούτω ώστε να διερευνήσουμε τον ευσταθή, το περιεχόμενο της πράξης κατ' εξουσιοδότηση και έχοντας γνώση της κατάστασης, ο εισηγητή θα μπορέσει να μοιραστεί και τις γνώσεις την, που έχουμε για το θέμα αυτό ε, με την Επιτροπή ΑΦΕΤ, Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτά αποφάσισαν οι και τώρα οι συνεισηγητές μας κατέθεσαν τα σχέδια έκθεσής τους για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά τις εκλογές. Η κυρία Ιζαμπέλ Τομά και ο Γιάν Ολμπρίχτ, οι συνεισηγητές μας, λαμβάνουν ήδη τις ευχαριστίες μας για την ποιότητα της εργασίας τους που αντανακλάται στο σχέδιο έκθεση που κατέθεσαν. Ποιος θέλει το λόγο? Ο Γιάννη Όλμπριχ θα αρχίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα κάνουμε από κοινού την παρουσίαση εγώ και η κυρία Τόμα. διότι έχουμε αναλάβει ο καθένας σε διαφορετικό κομμάτι της έκθεσης πρωτοβουλίας μας. Ε, να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με την ομοθεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να παρουσιάσει την ενδιάμεση αναθεώρηση το αργότερο στο τέλος του 2016. Και βέβαια η ενδιάμεση επανεξέταση στόχο έχει να δείξει ποια είναι η κατάσταση των δημοσιονομικών προοπτικών, αλλά καλύπτει και οτιδήποτε συνδέεται με αυτές, δηλαδή όλες τις πολιτικές που χρηματοδοτούνται από το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει το έγγραφο που θα δείχνει τι συμβαίνει σε όλες τις βασικές πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ψηφιστεί από το ε, Συμβούλιο η έκθεση αυτή. Ε, η δική μας αρμοδιότητα σύμφωνα με την ε, συνθήκη δεν είναι πολύ ευρεία. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το θέμα και γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε διαδικασία στην Επιτροπή μας με μια έκθεση πρωτοβουλίας. Να σας θυμίσω ότι στην ισχύουσα νομοθεσία λέει ότι μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση, εάν είναι απαραίτητο, εφόσον ενδείκνεται, θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση, να γίνουν διορθώσεις δηλαδή, τροποποιήσεις, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό, ως εισηγητές, προτείνουμε να συζητήσουμε την αναθεώρηση με τέτοιο τρόπο, ε, ώστε να ακολουθεί το έγγραφο που θα είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει με το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, τι είναι η επανεξέταση και τι είναι η αναθεώρηση. Η αναθεώρηση αφορά το δεύτερο μισό του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Πρώτα λοιπόν έχουμε την επανεξέταση, δεύτερον το τι θα πρέπει να αλλάξει και τρίτον ε, τι θα ισχύει μετά το 2020. Θα ήθελα εκ μέρους και των δυο μας να πω ότι δεν είμαστε ε, δογματικοί. Δεν λέμε ότι θέλουμε αναθεώρηση ήδη από την αρχή. Μετά όμως από όλες ε, τις συναντήσεις που είχαμε, τις ομάδες παρακολούθησης, τις ακροάσεις, συμπεριλαμβανομένης ε, της ακρόασεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα, το συμπέρασμά μας το οποίο παρουσιάζουμε στην έκθεσή μας είναι ότι το εφόσον ενδείχνεται το as appropriate είναι απολύτως σωστό διότι πιστεύουμε ότι στο δεύτερο μισό θα πρέπει επιγόντως να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και διορθώσεις στον ίδιο τον προϋπολογισμό, στην δομή του, στους μηχανισμούς του αλλά και στα νομοθετικά έγγραφα που συνδέονται με τον προπολογισμό. Και επιμένουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε, πρέπει οι τροποποίησεις αυτές να γίνουν επιγόντως. Έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας, μια τετριατία, 2017 έως 2020. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2021 για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές. Ταυτόχρονα παρατηρούμε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο την τάση να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο μετά το 2020. Αυτό κατά τη γνώμη μας αποτελεί μόνο μέρος του προβλήματος. Το άλλο μέρος του προβλήματος ε, είναι το δεύτερο μισό της παρούσας περίοδου. Επίσης, υπάρχει η τάση όταν κάτι δεν, τα δεν πάει πολύ καλά να λέμε ότι αυτό θα λυθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Όλοι μιλάνε λοιπόν για την ενδιάμεση αναθεώρηση, κανείς όμως δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Αυτό σημαίνει τι, ότι θα το συζητήσουμε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέταση χωρίς να αλλάξουμε κάτι. Εμείς ως εισηγητές προτείνουμε να γίνουν συγκεκριμένε τροποποιήσεις και διορθώσει. Και γι' αυτό Επιτρέψτε μου να σας πω ότι προτείνουμε η ε, ε, έκθεση πρωτοβουλίας αυτής ε, που είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι η έναξη της δημόσιας συζήτησης. Είναι λοιπόν το πρώτο βήμα που προτείνουμε και έτσι ξεκινάει η συζήτηση διότι μετά την ψηφοφορία του Ιουλίου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι απλά να περιμένει τα έγγραφα της Κομισιόν θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε μέχρι το τέλος της όλης διαδικασίας. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική μας θέση και μία τελευταία παρατήρηση για το πρώτο αυτό μέρος. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουμε αναπτύξει επαρκώς, διότι νομίζουμε ότι αυτό θα γίνει από τις ε, επί της αρμόδιες επιτροπές. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον πολιτισμό ή την εσωτερική πολιτική, διότι Πιστεύουμε ότι αυτά τα θέματα αποτελούν αρμοδιότητα των ε, διαφόρων επιτροπών και περιμένουμε τις δικές τους νομοδοτήσεις και ε, τροπολογίες. Δεν πιστεύουμε ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα πρέπει ε, να κάνει τη δουλειά των άλλων επιτροπών. Να μην σας εκπλήξει λοιπόν ότι κάποια στοιχεία απλά επισημένονται χωρίς να τα αναπτύξουμε σε βάθος. Όσον αφορά λοιπόν ε, την κατάσταση τώρα και την επανεξέταση, θα παρακαλούσα την κυρία Τομά να συνεχίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο συνεισηγητής μου, κύριο Όλμπριθ, ο στόχος μας ήταν να προσπαθήσουμε να εργαστούμε χωρίς προκαταλήψεις, αλλά έχουμε και κάποιες προαισθήσεις για το τι μπορεί να προκύψει από αυτή την κατάσταση. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια απεικόνηση της κατάστασης του προϋπολογισμού στο δυνατόν πιο αντικειμενικά και βάσει του άρθρου 2 προσπαθήσαμε κατά κάποιο τρόπο να συγκρίνουμε την αρχική πρόταση για το δημοσιονομικό πλαίσιο και συγχρόνως να δούμε τα τρία χρόνια που έχουν περάσει και το χρόνο που είναι εν εξελίξη, ποια ήταν, ποιος ήταν ο συσχετισμός μεταξύ του δημοσιονομικού πλαισίου και της λειτουργίας του προϋπολογισμού. Προχωρήσαμε λοιπόν φάκελο με φάκελο. Είδαμε ότι είχαμε σημαντικά προβλήματα προϋπολογισμού. Φυσικά, σε ό,τι αφορά την έκταση των προβλημάτων Ξεκινήσαμε με την προσφυγική κρίση, όπως λέγεται, αλλά μάλλον πρέπει να μιλάμε για, ένα φαινόμενο μετανάστευσης, κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφτεί βέβαια στην, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το 2014, 2015 αλλά ιδίως 2016 οδήγησε σε σημαντικά ποσά του προϋπολογισμού με την υπέρβαση των οροφών κατά 1,5 δισεκατομμύριο στην κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά την ε, υποδοχή των μεταναστών αλλά και την ασφάλεια των συνόρων, τη Frontex κτλ. Είδαμε επίση ότι έχει τέθει σε εφαρμογή ένα νέο μηχανισμό ανθρωπιστικού χαρακτήρα, έκτακτη ανθρωπιστική αρρωγή, ο οποίο μέχρι τώρα αφορούσε μόνο χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη φορά χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί για την Ελλάδα. Στην κατηγορία 4 έχουμε επίσης υπέρβαση των οροφών, μικρότερη από την κατηγορία 3 βέβαια, <clears throat> αλλά έχει γίνει κάτι το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στην Επιτροπή μας, να δημιουργούνται εξωτερικά καταπιστεύματα. Εκτός λοιπόν της δυνατότητας να λειτουργήσει ο έλεγχος της Επιτροπής μας μέσα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσιολογικά θα έπρεπε και αυτά τα καταπιστέγματα να ενσωματωθούν μέσα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς υπάρχει η κρίση επενδύσεων η οποία δεν είχε οδηγήσει σε συγκεκριμένα μέτρα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά μετά από τις εκλογές του 2014 και την έλευση της νέας Κομισιόν έλαβαν χώρα αποφάσεις για να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την παινία επενδύσεων με το λεγόμενο σχέδιο Juncker και το οποίο χρησιμοποίησε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή εγγυήσεων και περιόρισε <clears throat> δύο από τις πιο ελπιδοφόρες στον τομέα των επενδύσεων θέσεις του προϋπολογισμού, γιατί η έρευνα, η δημιουργία υποδομών, σύνδεσης και μεταφορών θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι είναι οι μελλοντικέ επενδύσεις. Τουλάχιστον για την έρευνα αυτό είναι σίγουρο. Αυτές οι δύο γραμμές του προϋπολογισμού λοιπόν ακροτηριάστηκαν σε μια κατάσταση που ήδη είχαμε προβλήματα για τον προϋπολογισμό και κάτι ακόμα το οποίο δεν πρέπει να λησμονήσω πρέπει να αναφερθώ και στη διαπίστωση που έχουμε προβεί σε αυτήν εδώ και πολύ, πολλά χρόνια ως Επιτροπή Προεπολογισμών τη λεγόμενη κρίση των πληρωμών, των ποσών προς εκταμίευση, των ΡΑΛ. Από το 2010-2011 δεν έχει σταματήσει η αύξηση αυτών των ποσών προς εκταμίευση και ακόμα και όταν ξεκινάνε τα πολιετή προγράμματα είναι μια εποχή που μπορεί κανείς να απορροφήσει κάποιους λογαριασμούς γιατί εκείνουν τα προγράμματα βραδέως. Όταν αρχίζουν και συσσωρεύονται οι αιτήσει πληρωμών θα είμαστε και πάλι αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχει γιατί δεν το επιτρέπουν ποτέ οι συνθήκες να υπάρχει ένα συνεχιζόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού το οποίο μάλιστα και διονγκώνεται. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο της αύξησης των δαπανών που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των συνόρων, με την υποδοχή των προσφύγων, με, τις, ε, με το πρόγραμμα Juncker επενδύσεων και επίσης έχουμε και την πρωτοβουλία για τους νέους που είχε προγραμματιστεί για δύο χρόνια μετά. Το πρόγραμμα αυτό δεν είχε θεσπιστεί για το χρονικό διάστημα 2016-2020, γιατί περιμένουμε από το 2016 όταν μπορέσουμε να δώσουμε και πάλι χρηματοδότηση σε αυτό το πρόγραμμα. Δυστυχώ τώρα η κατάσταση τη απασχόληση των νέων δεν έχει βελτιωθεί καθόλου, αλλά το 2016 δεν είναι ένα έτος το οποίο να προβλέπει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων. Έχουμε επίσης και τα στοιχεία της ευελιξίας στο αποθεματικό για απρόπτα, στο μέσο ευελιξίας, στην χρησιμοποίηση των περιθωρίων που χρησιμοποιήθηκαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και βέβαια χρησιμοποιήθηκαν πλήρως, ενώ δεν έχουμε διανύσει ούτε το μισό της πολυεκτικούς ε, περίοδους και επομένως τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε μία περισσότερο ανάσα σε επίπεδο προπολογισμού. Αυτά θέλω να σας πω λοιπόν. Και τώρα μετά από την λεπτομερή και δελεχή εξέταση όλων των θέσεων του προϋπολογισμού το χρονικό διάστημα 14-15 και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό για το 2016 βλέπουμε να υπάρχει μια σημαντική απόκληση μεταξύ αυτού που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και τις προτεραιότητες. Με το πρόσθετο πρόβλημα ότι οι νέες προτεραιότητες στον προπολογισμό <clears throat> δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις προηγούμενες. Δεν βλέπουμε ούτε μείωση της ανεργίας των νέων, ούτε αύξηση του προπολογισμού. Αυτή η απόκληση λοιπόν που παρατηρείται στον προπολογισμό, αν τηρήσουμε το άρθρο 2, μας οδηγεί μαθηματικά στην ανάγκη μιας αναθεώρησης του, των δημοσιονομικών πρόπτικων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η τροποποίηση. είμαι περιορισμένος σε σχέση με τον αριθμό σελίδων που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτή την έκθεση, αλλά νομίζω ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι ζητούμε να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ήδη για το 2017 έναντι του πλαισίου που είχε προβλεφθεί. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει. Ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστούμε Ιζαμπέλ Τομα. Ε, συγγνώμη διακόπτει ο κύριος Ολμπρίχτ αλλά δεν τελειώσαμε. Έχουμε και άλλα δύο τμήματα. Ένα θα πω εγώ, ένα η κυρία Τομα. Μπορείτε να το διαβάσετε το κείμενο, οπότε θα συνοψίσουμε. Εάν το συμπέρασμα είναι ότι χρειαζόμαστε αναθεώρηση, λέει μες στο τρίτο τμήμα της έκθεσης τι κατά τη γνώμη μας πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί. για τις ε, δεσμεύσεις υποχρεώσεων. Α, και υπάρχει και το πρόβλημα της επιστροφής των κονδυλίων που έχουν ε, χρησιμοποιηθεί για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Η εγγύηση για την νεολαία που εκπνέει. Το αναφέραμε ήδη αυτό. Για τα τμήματα 3 και 4 επίσης, ε, πάλι για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Για τις πιστώσεις πληρωμών, τώρα, θέλουμε να αποφύγουμε και πάλι μια κρίση πληρωμών. Και τι είναι αναπόφευκτο. Τα πλαφόντα, τα όρια. αυτό το επίπεδο πληρωμών ε, θα μας οδηγήσει πάλι σε δυσχερέστατη θέση. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Έχουμε και την ε, αδύνατη αποστολή που θα να εκπληρώσουμε, δηλαδή ό,τι σχετίζεται με το πλάνο να μένει στο προϋπολογισμό. Επικίνδυνη και αδύνατη αποστολή. Θα είναι ε, πολύ ισχυρέ οι αντιδράσεις. Το πλάνο πρέπει να μείνει στον προϋπολογισμό. Επίσης, ε, θέμα ευελιξίας για τα όρια και για το χρονοδιάγραμμα. Εμείς προτείνουμε αλλαγές, διότι προς το παρόν δεν έχουμε καμία ευελιξία στο πολιετές. Αυτό το εξηγούμε και στον προϋπολογισμό. Με ποιο τρόπο θέλουμε να αλλάξουν οι κανόνες. Επίσης, ε, η απλούστευση και τα χρηματοδοτικά μέσα. Θέλουμε πραγματικά να υπάρχει σοβαρή απλούστευση, όχι συμβολική εξοραϊστική, διότι είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα σήμερα. Πιστεύουμε ότι τώρα πρέπει να απλουστευτεί το σύστημα και ο δημοσιονομικός κανονισμός, το ίδιο ε, και το CPR. Πρέπει να δείξουμε πολιτική βούληση. Ε, να δείξουμε ότι θέλουμε να συμβάλλουμε στην απλούστευση, τροποποίηση και απλούστευση του κανονισμού. Για το νόμο για, για το Ταμείο Συνοχή, παραδείγματο χάρη, τι, ποιο είναι το πρόβλημα με την νομοθεσία. Είναι κανονιστικό το ζήτημα, είναι υπερβολικά περίπλοκο το σύστημα. Εάν ναι, ταχύτερο δυνατόν να το απλουστεύσουμε. Αλλά όχι τώρα, αλλά ούτε και να τα αναβάλουμε μετά το 2020. Αυτό είναι το πρόβλημα γενικά τι γίνεται με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Τώρα, ποια απλούστευση πρέπει να κάνουμε. για το πλεόνασμα. Τώρα θα πρέπει να ε, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Ε, μιλάμε λοιπόν για το δεύτερο ημιζή του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και τώρα μετά την αναθεώρηση το 2020 θα έχουμε το δεύτερο τμήμα. Oui, effectivement, euh, nous nous sommes dit que euh, nous ne pourrions pas... Πράγματι, είπαμε, είχαμε πει ότι πρέπει να τα ρυθμίσουμε όλα όταν θα γινόταν η αναθεώρηση. Ήμασταν φιλόδοξοι σε σχέση με την αναθεώρηση, αλλά ορισμένα από τα θέματα της αναθεώρησης θα πρέπει να τύχουν μια πιο ενδελεχούς συζήτηση για την αναθεώρηση. Εν είπαμε ότι τα θέματα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και προτείναμε συγκεκριμένα. πολλές πτυχές, πρώτη των οποίων είναι αυτή τη διάρκεια γιατί αυτό ήταν κάτι το αμφιλεγόμενο, θυμόσαστε, όταν έγινε διαπραγμάτευση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το γεγονός ότι η διάρκεια του είναι αποσυνδεδεμένη από την, από την διάρκεια της θητείας της Κομισιόν και θέλουμε να επανέλθουμε στη λογική μιας διάρκειας πέντε ετών που ανταποκρίνεται στο, στη δημοκρατική εντολή του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και συγχρόνως για μακροχρόνια ορατότητα του προϋπολογισμού προτείνουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο 5 συν 5 ίσον 10 σε ό,τι αφορά για την πολιτική συνοχή, για τις επενδύσεις, για τις μακροχρόνιες ενέργειες. Πρέπει λοιπόν να <clears throat> κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των θεμάτων πρέπει να τύχουν ορατότητα. 5 συν 5 λοιπόν και αυτών που συνδέονται με μια συγκεκριμένη πολιτική εντολή 5 χρόνια μονάχα. Αναφέραμε και κάποιες ε, αρχές οι οποίες φαίνεται ότι έχουν περάσει στα ύδατα της στιγός. Καταρχήν πρέπει να είναι ενιαίος ο προϋπολογισμός, να υπάρξει ενότητα του προπολογισμού. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν όλα αυτά τα καταπιστεύματα, όλα αυτά τα εξωτερικά ταμεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπόκειται στην ίδια διαδικασία ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είχαμε υπενθυμίσει την αρχή της ισορροπίας, η οποία με την κρίση των πληρωμών ουσιαστικά και αυτό έχει <clears throat> λησμονηθεί την οικουμενικότητα του προϋπολογισμού, γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο υπάρχουν κονδύλια τα οποία προσδιορίζονται για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καταρχήν η αρχή της οικουμενικότητας του προϋπολογισμού επιτρέπει την ετήσια προσαρμογή ή την αρχή της διαφάνειας κτλ. Όλες αυτές οι αρχές λοιπόν πρέπει να επενδυμιστούν, αλλά έχουμε επιπλέον διαπιστώσει και προτείνουμε εδώ να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός για νέα εργαλεία <clears throat> ευελιξίας, γιατί θεωρούμε ότι αυτά που έχουμε τώρα δεν ήταν προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, η ανθρωπιστική βοήθεια η οποία αφορούσε μονάχα τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες, οι περιορισμοί, για την ε, χρήση αυτών των κονδυλίων, η ανάγκη επιστροφής κονδυλίων κτλ. Προτείνουμε λοιπόν και αυτό το θέμα να επανεξεταστεί τα εργαλεία ευκαμψίας ώστε να μπορούν να είναι πιο εύχριστα και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μας λέει ότι η διευκόλυνση για την Τουρκία πρέπει να είναι πιο εύκαμπτη. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα αυτή η απαραίτητη ευκαμψία. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία των προτάσεών μας. Και φυσικά υπάρχει πίσω από αυτά η θέληση, όπως είπε και ο κ. Όλμπριχτ, η θέλησή μας να υπάρξει μια αναθεώρηση επειδή είναι απαραίτητη και να μην καταλήξουμε να πέσουμε στην παγίδα που να μας πούν ότι δεν έχει νόημα να αλλάξουμε τώρα, γιατί ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2017 θα αρχίσουμε συζητήσεις για ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτε πρέπει να πέσουμε στην αντίστροφη παγίδα να φτιάξουμε ουσιαστικά ένα αυτοσχέδιο προϋπολογισμό αναθεωρημένο για το δεύτερο μισό του τωρινού πλαισίου και να αφήσουμε για τις ελληνικές καλένδες την συζήτηση για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε και αναθεώρηση και προετοιμασία του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και το νέο αυτό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ε, άνοδο των οροφών και θα απαιτήσει να υπάρχουν νέοι πόροι. Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί απλώς να ζητήσει περισσότερα χρήματα από τα κράτη-μέλη χωρίς να σκεφτεί και σοβαρά για τους πόρους, για τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία μπορούν να εξευρεθούν αυτοί οι πόροι. <clears throat> Αυτά λοιπόν είναι και το βασικό στοιχείο στην έκθεση μας στο τέλος που λέμε ότι το θέμα των ιδιών πόρων που είχε τεθεί ήδη όταν γινόταν διαπραγμάτευση το 2013 για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το θέμα των ιδιών πόρων είναι ένα διαρθρωτικό στοιχείο και ένα δομικό στοιχείο χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική μεταρρύθμιση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, ούτε μπορεί να υπάρξει φιλοδοξία για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο γιατί είναι αξιοθαύμαστη δουλειά που κάνατε Ε, θέλω να τονίσω ότι πραγματικά είναι αξιέπαινος ε, ο ενθουσιασμός που δείχνετε και ο ζήλος σας δεδομένων και των προβλημάτων ε, που εγγράφονται στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει ελοχεύει ο κίνδυνος πάντοτε πιθανών απογοητεύσεων στο, σε σχέση με τις φιλοδοξίες σας, αλλά σε κάθε περίπτωση την κάνετε την προσπάθεια και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής μας. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ε, παρεμβάσεων. ο Φερνάντες θα πάρει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους συνεισηγητές. Είναι εξαιρετικά ποιοτική η δουλειά που έκαναν και υψηλή η φιλοδοξία τους είπατε εσείς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο ρεαλισμός τους που χαρακτηρίζει αυτή την έκθεση διότι εντοπίζει τις ανάγκες ε, που έχουμε και ε, τις ανησυχίες που πρέπει όλοι να συμμεριζόμαστε. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εξή. Εμεί χρειαζόμαστε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε αξιολόγηση του πολιτού δημοσιομικού πλαισίου. Όποιο το αρνείται αυτό, ε, αρνείται και την πραγματικότητα. Ε, χρησιμοποίησαμε τη μέγιστη διαθέσιμη ευελιξία στον προπολογισμό το 2016, ε, πάρα από 1,5 δι. Ε, στο μέσο ευελιξίας. Ε, χρησιμοποιήσαμε το Ταμείο για την ε, Αφρική, το Ταμείο για την Υποστήριξη των Προσφύγων στην Τουρκία, το νέο Ταμείο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη αξιολόγησης ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και ελπίζω να αναγνωρίσει το αυτονόητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, να μην αρνηθεί, να μην κλείσει τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα το Συμβούλιο. Αυτό θα ήταν ένα θετικό μήνυμα. Τούτου λεχθέντος θεωρώ ότι όπως ανέφεραν και οι συνεισηγητές είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία αλλά δεν μπορεί να έχουμε μειώσεις, περικοπές στον προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε ε, να βάλουμε αυτά τα νέα ε, ταμεία και τα trust funds μέσα στον προϋπολογισμό αλλά όχι από την άλλη να περικόπτουμε τις ε, δαπάνες του προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε να έχουμε ανώτατο όριο το 1% στον προϋπολογισμό και ταυτόχρονα να βάζουμε όλα τα ταμεία να τα εντάσσουμε προσθέσουμε στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι de facto περικόπτουμε τον προπολογισμό με αυτόν τον τρόπο. Οπότε είναι απαραίτητη η ευελίξια. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ευελίξια όταν ενέκρινε το πολιετέ το Κοινοβούλιο και όταν τι απέτησε αυτέ τι προσαρμογέ ε, ε, με διορθωτικού προπολογισμού, δεν θα είχαμε ανταποκριθεί σε αυτέ τι ε, κατεπίγουσε ανάγκε που αντιμετωπίσαμε, παραδείγματο χάρη με το σχέδιο Juncker, με το Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων. Με αυτή την ευελιξία ακριβώς καταφέραμε ε, μέσα από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα που έχουμε. Αυτή η ευελιξία όμως προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείται εις το έπακρον και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει πώς γίνεται οι κυρώσει που είναι πόροι του προϋπολογισμού δεν προστίθενται στον προϋπολογισμό αλλά επιστρέφουν όλα τα πρόστιμα, όλες οι κυρώσει ε, στα, στα κράτη-μέλη όπως ε, ε, δείχνει και η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα ποσά πρέπει να επανεγράφονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν αυτού και πέραν των προϋπολογισμών των δεν πρέπει να χάνουμε κονδύλια ε, από τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Πρέπει να μετατρέπονται όλες οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε πιστώσεις πληρωμών. Δεν μπορούμε να χάνουμε κονδύλια με αυτόν τον τρόπο. Για τη διάρκεια, συμφωνούμε όλοι πως υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση και το ιδανικό θα ήταν η εντολή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αυτή η πενταετή σε περίοδο να συμπίπτει χρονικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως ποτέ δεν καταφέραμε να υπάρξει αυτή η χρονική σύμπτωση. Και Ενάμιση χρόνο ε, στην καλύτερα των περιπτώσεων διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, συνήθως πολύ περισσότερο από αυτό. Με τόσο μακρές διαπραγματεύσεις ποτέ δεν θα καταφέρουμε να υπάρξει χρονική σύμπτωση με αυτή την ε, πενταετή περίοδο. Αφήστε που έχουμε και πολιτικές, προκειμένου πολιτική της συνοχής, που έχει αυτό τον κανόνα, νη συν τρία. Ε, και τα κράτη-μέλη αποφάσισαν αυτό τον κανόνα, νη συν τρία. Και άρα με τα πέντε χρόνια, με την πενταετή περίοδο, ποτέ δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε, ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε σύμπτωση λόγω αυτού του κανόνα. Θα ήθελα να ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύει ε, σε σχέση με την ε, αναθεώρηση. ακολουθεί τη γραμμή που εισηγούμαστε εμείς και πότε θα καταθέσει την πρόταση για την αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν συμφωνήσει θα πρέπει να καταθέσει την πρόταση για να μπορέσουμε πολύ απλά και το ξαναλέω να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Μανκά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο συγητές. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό το έργο και των δύο, όπως είπε και ο κύριος Φερνάντης προηγουμένως. Ίσως είναι ιδεαλιστική προσέγγιση σας, αλλά αν μπορέσετε να πείσετε για αυτή την κατεύθυνση, τότε τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν. Συμφωνώ με τον κύριο Όλμπριχτ ότι είναι δύσκολο να παραμένουν πλεονάσματα από τον προϋπολογισμό που γυρίζουν στα κράτη-μέλη, γιατί το κάθε κράτος προσπαθεί να πάρει αυτά τα χρήματα πίσω. Είναι καλύτερα να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα από τους ε, ίδιους πόρους. Τότε δεν θα μπορούν αυτά τα κονδύλια να χάνονται από τον προϋπολογισμό. Κάνετε μια πολύ καλή ανάλυση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλος ο κόσμος. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό γίνεται σαφές ότι συσσωρεύονται όλα τα στραβά την ίδια στιγμή. Δηλαδή όλες οι αναποδίες, η ανεργία των νέων, η κρίση προσφυγική, η οικονομική δυσπραγία, όλα αυτά έχουν το αποτέλεσμα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους που θα μπορούσαμε να βρούμε για να βελτιωθούν τα πράγματα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό και αντίστοιχα ταμεία μπορούν να βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την φορολογική, την φοροαποφυγή. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να κάνει όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα ώστε ο πληθωρισμός να μείνει μικρός. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να χρηματοδοτήσει με τέτοιο τρόπο το τραπεζικό σύστημα ώστε να, να ενταθεί η να ενταθούν οι επενδύσεις στα θέματα της, ε, κλιματικής, ενεργειακής απόδοσης κτλ. Ο κύριος Δράγκη είπε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο, αλλά εδώ η ιδέα αυτή είναι ενδιαφέρουσα, θα έπρεπε να το εξετάσουμε και στην Επιτροπή μας, να δούμε με ποιο τρόπο τα χρήματα της ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να χρηματοδοτούν τις πιο σημαντικές στρατηγικές. Αν οι στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τα απαραίτητα ε, μέσα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Χρειαζόμαστε πρόσθετα χρήματα για την, για Τουρκία και άλλες τέτοιες πολιτικές. Επομένως, η δική μου αίτηση είναι ας χρησιμοποιήσουμε με πιο στοχευμένο τρόπο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να καλυφθούν οι κυρίες προτεραιότητες μου. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Λεβεντόφσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συντάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε που ευθυγραμμίζεται λίγο πολύ με τα όσα είπαν η κυρία Τόμα και ο κύριος Όλπριχτε. Βλέπουμε ένα πολύ ισχυρό πνεύμα συνεργασίας ε, από πλευράς των συνεισηγητών, το οποίο είναι πολύ θετικό. Όσον αφορά τον δημοσιονομικό προϋπολογισμό, θυμάμαι ε, τον τελευταίο γύρο συζητήσεων. Ε, πάντα είναι χαρά μου να συνεργάζομαι, αλλά απέτησε πολύ χρόνο, κάτι που δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό όσον αφορά τις μελλοντικές προσπάθειες. Ε, ως συντάκτης της Επιτροπής Ήτρε όμως ε, πρέπει να σκεφτεί κανείς τις ευαισθησίες της Επιτροπής Ήτρε. Αλλά αυτό που το, το κυριότερο που λέμε είναι ότι ζητάμε αναθεώρηση και όχι απλά επανεξέταση. Και επίσης θα πρέπει να αποκατασταθούν ε, τα, οι, πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατικών Επενδύσεων, κάτι που είναι αδύνατο να γίνει αν δεν γίνει πραγματική αναθεώρηση ε, του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρει την Επιτροπή Ήτρε το πρόγραμμα Horizon 2020, τον Καλλιλέο για παράδειγμα, ε, είναι από απολύτως ε, χρήσιμο και επίκαιρο ε, πρόγραμμα. Ε, το κομμάτι αυτό του προπολογισμού λοιπόν έχει να κάνει κυρίως με το μέλλον και επίσης μία μικρή προειδοποίηση όσον αφορά την εφαρμογή. Η αναθεώρηση που θα σχετίζεται με την εφαρμογή ακούγεται ε, σαν να είναι αυτονόητο, αλλά είναι πολύ νωρίς για να δούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί ε, στο πλαίσιο του παρόντος ε, πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει λοιπόν να σας προειδοποιήσω να μην κάνουμε πολλές αλλαγές με βάση του τι έχει γίνει μέχρι τώρα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστέρηση σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές, αλλά ιδίως θέλω να τους συγχαρώ απόλυτα, γιατί έχουν κάνει ένα έργο το οποίο ήταν πάρα πολύ εξισορροπημένο, πολύ λογικό, πολύ καλοφτιαγμένο. Δεν ξέρω τώρα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να το πάρει αυτό το έγγραφο και να το παρουσιάσει σχεδόν σαν μια ανακοίνωση της Κομισιόν γιατί είναι η καλύτερη βάση για μια αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, όχι προτάσεις, προτάσεις που στρέφονται προς το μέλλον. Είναι πάρα πολύ καλή η εργασία των δύο εισηγητών. Και νομίζω ότι βρήκανε το μέσο δρόμο <clears throat> μεταξύ των ε, προτάσεων που έχουν διατυπωθεί. Υπάρχουν ε, οι, τα σημεία που πρέπει να αλλάξουν τώρα μέσα στο το τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο. Συγχρόνως όμως πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει και το 2020 και επέκεινα. Εκεί τρέφω ένα φόβο ότι ενδεχομένως αυτές οι προτάσει για τους ίδιους πόρους, για τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου δεν πρέπει να μας αφαιρέσουν την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τώρα τις αλλαγές που χρειάζονται. Το είπε ο κ. Φερνάντες, είναι φιλόδοξες οι προτάσει του, αλλά είναι και ρεαλιστικές, συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Αυτό που καταδεικνύει η έκθεση αυτή είναι ότι υπάρχει μια απόλυτη αδύρυτη ανάγκη να τροποποιηθεί το πλαίσιο και ορισμένε πολιτικές μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί αλλιώς θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε επίπεδο πραγματικότητας. Όταν εμείς είχαμε εγκρίνει στην προηγούμενη θητεία αυτό το πλαίσιο, το δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τονίσει ιδιαίτερα την ύπαρξη αυτού του άρθρου για την αναθεώρηση στα μέσα του δρόμου. Γιατί είχαμε τονίσει τότε ήδη ότι υπήρχαν προβλήματα στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέραμε ότι σίγουρα θα προκύψουν προβλήματα στις ε, πληρωμές. Ξέραμε ότι τα χρήματα για την εγγύηση για τους νέους δεν ήταν αρκετά και έπρεπε να αυξηθούν και όλα αυτά χωρίς να ξέρουμε ότι θα προκύψει και η κρίση των προσφύγων χωρίς να ξέρουμε ότι πρέπει ένα τμήμα της κατηγορίας 1α θα πρέπει να αναδιαρθωθεί για τη χρηματοδότηση του σχεδίου Juncker. Ξέραμε ήδη τότε ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση και τώρα έχουμε συσσωρεύσει πολύ περισσότερα επιχειρήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να τα τονίσουμε αυτά τα σημεία τα συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα την ευελιξία, γιατί είδαμε πόσο σημαντικό ήταν να μπορούμε να έχουμε κάποια ευελιξία αλλά συγχρόνως και επειδή είναι σαφές ότι η ευελιξία που έχουμε ενώπιον των προκλήσεων που θα έχουμε μέχρι το 2020 είναι ανεπαρκής και επίσης πρέπει να τονίσουμε την απλοποίηση. Μιλώ για μια απλοποίηση, γιατί κάθε φορά που αλλάζουμε κάτι το κάνουμε πιο πολύπλοκο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε πιο πολύπλοκα τα πράγματα, γι' αυτό ίσως πρέπει να αρχίσουμε να τα απλοποιούμε. Αλλά αν δεν μπορούμε να έχουμε τα μία για την εγγύηση για τους νέους που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επειδή είναι υπερπολύπλοκος ο κανονισμός. Και το ίδιο με, την, με αρρωγές προς τη γεωργία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι τόσο πολύπλοκος ο κανονισμός τους που δεν ξέρουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία να απλοποιήσουμε όλους τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις που έχουμε θεσπίσει. Ο Κάροντι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους ε, εισηγητές ε, για την ε, πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει για το πολιτικές δημοσιονομικό πλαίσιο και για το πού βρισκόμαστε. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την προσφυγική κρίση διότι ε, έτσι φαίνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο ότι πρέπει να έχουμε αναθεώρηση του πολιετού σε δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, έχουμε ε, μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση εν εξελίξη και εντός των συνόρων και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μέχρι στιγμής. Επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Λεβαντόφσκι είναι απολύτως απαραίτητο να προστατεύσουμε κονδύλια όπως είναι αυτά του ορίζον 2020 και της διευκόλυνσης σε συνδέοντας, της Ευρώπης, ε, συνδέοντας την Ευρώπη. Δεν έχει νόημα να αφαιρούμε χρήματα από μια βέβαιη επένδυση για το μέλλον μας ε, και να τα διαθέτουμε σε μια βέβαιη επένδυση που μπορεί να είναι επιτυχής αλλά είναι πολύ διαφορετική από αυτήν για την οποία προορίζονταν αρχικά τα κονδύλια. Και ε, επίσης ε, κάτι που μάλλον δεν θα εκπλήξει πάρα πολύ τους συναδέλφους, η επόμενη μου παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει καταρχάς να εξετάσουμε τους υπάρχοντες πόρους και το πώς μπορούν να αναδιανεμηθούν για να πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης, θα ήθελα να σας καλέσω να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά ε, το 5 συν 5 όσον αφορά την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, υπάρχει ο φόβος να καταλήξουμε σε δεκαετή προγράμματα με ενδιάμεση αναθεώρηση. Και άλλωστε μέρος της επιτυχίας ήταν ότι είχαμε τα επταετή προγράμματα όπου μπορούσε να παρέμβει το Κοινοβούλιο. Υπήρχε έτσι κάποιο είδος σταθερότητας και φοβάμαι Νομίζω ότι έτσι θα χάσουμε την σταθερότητα μακροπρόθεσμα και πάλι θα ήθελα να τονίσω ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά οι συνεισήγητες. σε ευχαριστούμε. Ο Ζεράν Ντεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τη σειρά μου να επενέσω και εγώ τους συνεισηγητές. Ε, πραγματικά, ε, όχι μόνο με ικανοποίησε αυτό το έγγραφο, ήταν και ευχαρίστηση ε, να, το, όταν το διάβαζα, διότι είναι ξεκάθαρη, σαφέστατη η επιχειρηματολογία και ε, η κυρία Τομά έχει πραγματικά μεγάλες φιλοδοξίες, τις οποίες εγώ συμμερίζομαι. Είναι απαραίτητη να μείνει η εξελόγηση, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα είναι εύκολη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να στοχεύσουμε καλύτερα. Ποια είναι τα βασικά στιγμία. Πρώτον, ε, είναι ανησυχητικοί οι προπολογισμοί σε διάφορα κράτη-μέλη, το ίδιο και η πολιτική κατάσταση. Είναι και χειρότερη, μπορώ να σας πω, ή ε, πολύ πολύ σύντομα να συμβεί κάτι τέτοιο, αν παρακολουθήσετε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις σε κάποια κράτη-μέλη. Τούτου με μεγάλη ακρίβεια, σαφήνεια και διάβια ε, εντόπισαν οι συνεισηγητές τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Έξι θα αναφέρω, μεταναστευτική κρίση, προσφυγική, ε, χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, ανάγκη στήριξη των μικρομεσαίων, ε, απασχόληση για τους νέους, ε, εσωτερική ασφάλεια, προβλήματα γεωργίας και δυσκολίες ε, ή πώς να πω ε, δράμα, εν πάση περιπτώσει η κατάσταση με τις ε, πληρωμές στον προϋπολογισμό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία και συμφωνούμε με την ανάλυση που κάνουν και τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Βεβαίω, θα ήθελα ε, ελαφρώς να τροποποιήσω κάποιες από τις προτάσεις που κάνουν. Για τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας ε, και την ε, προσφυγική δεν επαρκεί το ε, όριο του τμήματος 3. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Επίσης είναι ε, τραγικές εξελίξεις σε κάποια κράτη-μέλη και ακόμη και για ανθρωπιστικούς λόγους θα χρειαστούν ε, παρεμβάσεις που επισύρουν χρήση πολύ υψηλότερων κονδυλίων. Μήπως πρέπει να μιλήσουμε για το τμήμα 1, διότι ε, θέλουμε να έχουμε τις δεσμεύσεις για το ΕΦΣΙ από τη μία, από την άλλη όμως να διατηρήσουμε τις δυνατότητες που δίνει το ΕΦΣΙ για τις επενδύσεις και για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Όλμπιχ με κοιτάει καλά-καλά. Δεν το είδα μέσα. Ίσως ε, δεν μου ξέφυγε διαβάζοντάς το. Δεν ξέρω αν το έχετε προτείνει. Ε, πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, για τις πληρωμές. Ζητάμε ένα πραγματικό σχέδιο πληρωμών. Μας την έχουν φέρει επανειλημμένα. Μας λένε αν θα κάνουμε. Τίποτα δεν γίνεται όμως. Κάθε φορά που έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει, μα μην ανησυχείτε του χρόνου, ε, θα εχουμε δύο, τρία, δις και κανένα πρόβλημα με τις πληρωμές και τελικά μεγαλώνει η χιονοστιβάδα και πάλι στο ίδιο σημείο θα, στην ίδια δύσκολη θέση θα περιέλθουμε. Λοιπόν, για τις πληρωμές ε, πρέπει ξεκάθαρα να αναφέρεται ε, και ενώ δεν ισχύει, μάλλον αναφέρεται στη Διοργανική Συμφωνία του Δευτέρας Δεκεμβρίου του 2013, δεν αρκεί αυτό, πρέπει να προβλέψουμε κάτι συγκεκριμένο ε, στα πλαίσια της ε, νέας αξιολόγησης και της νέας ε, τροποποίησης της Διοργανικής Συμφωνίας. Επίσης, προσοχή, γιατί έχουμε τα ειδικά χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία εντάσσονται στα όρια του προπολογισμού, εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι αποβαίνει αυτό εις βάρος του Κοινοβουλίου και θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μαζί σας και κάποιες ιδέες, κάτι που δεν αναφέρεται μέσα στο, στην έκθεση, για τη διατροφή, για τα μέσα ευελιξίας. Τα λέγαμε και την περασμένη φορά, θα καταθέσω συγκεκριμένε προτάσεις για να τις συζητήσουμε. Στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων νομίζω δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε ακόμη. Πρώτον, με τι συναρμόδιε επιτροπές να κάνουμε ε, όσο το δυνατόν ακριβέστερη αποτίμηση των συμπληρωματικών μα αναγκών για τα διάφορα τμήματα μέχρι ε, την εκπνοή του ε, ενισχύως δημοσιονομικού πλαισίου. Διότι είναι προφανείς αυτέ οι ανάγκες δεν μπορούμε ε, παρά να τις ικανοποιήσουμε και άρα θα πρέπει να γίνει ακριβής αποτίμησή τους. Επίσης για τη στρατηγική μας, ε, ποιο είναι το μίξε που θα προωθήσουμε για τη διεκδίκηση των αξιώσεων μας. Θα ρίξουμε το βάρος στην αύξηση των ορίων ή όπως ακούω ότι να οργιάζουν οι φήμες από το Συμβούλιο θα ε, δουλέψουμε τα μέσα ευελιξίας αύξηση αφενός του ρίου και αφετέρου πιο ευέλικτη ευέλικτους όρους εφαρμογής, παραδείγματος χάρη με ποιο τρόπο μπορούν να επιτευχθούν διαφορετικού είδους πλειοψηφίες ε, στο Συμβούλιο, δηλαδή αλλαγή ε, του τρόπου λήψης αποφάσεων βάσει πλειοψηφία στο Συμβούλιο Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να καταγράψουμε όλα αυτά τα στοιχεία συγκεκριμένα, όμως ε, από πλευρά στρατηγικής θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι ώστε να διαπραγματευόμαστε από θέση ισχύας. Και θα κλείσω τώρα, είναι αξιοθαύμαστο αυτό το έγγραφο πραγματικά και ε, ε, συναντιούνται τα μεγάλα πνεύματα, δύο μεγάλα πνεύματα και πραγματικά είναι αξιέπαινο το αποτέλεσμα. Ε, αλληλογονιμοποιούνται. Ο κύριος Μαραγκάλ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία συμμερίζομαι με τους προλαλήσαντες και είναι πολλά. Σίγουρα οι έπαινοι που διατυπώθηκαν για τους εισηγητές είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Αξίζουν κάθε έπαινο. Θέλω απλώς να διαφοροποιηθώ σε ορισμένα σημεία γιατί νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις στην έκθεση. Μπορούμε λοιπόν να συγκεκριμενοποιήσουμε ενδεχομένω καλύτερα την φιλοδοξία μας να υπενθυμίσω ποιο είναι το σημείο κίνησής μας. Εγώ δεν ήμουν εδώ όταν ξεκίνησε αυτή η, αυτό το εγχείρημα, αλλά αναφέρεται και στο πολιτές πλαίσιο 2014-2020 οι πράσινοι που εκπρόσωπο εδώ σήμερα ψήφισαν κατά της τελικής συμφωνίας για τους λόγους που τώρα αναδύονται ως επιχειρήματα υπέρ μιας πραγματικής αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό που δημιουργήθηκε το 2014-2020 ήταν πολύ σφιχτό, πολύ περιορισμένο, πολύ άκαμπτο, χωρίς καμία απόλυτη δέσμευση για αλλαγές και παραμένει η ανάγκη για μια μεταρρύθμιση των ιδιών πόρων που το είχαμε τόνισει πριν από δύο χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε λοιπόν όλα αυτά. πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε από κοινού στο πολιτικό πλαίσιο που ανοίγει η πρόταση των εισηγητών. Και αυτή τη φορά θα πρέπει να λειτουργήσουμε με την λογική να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα βασικά σημεία στη συμφωνία. Και θα το πράξω και εγώ από τη δική μου πλευρά με τις ε, τροπολογίες μου και φυσικά συμμεριζόμαι απόλυτα αυτά που είπαν οι συγητές ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια αυθεντική αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Δύο βασικά ερωτήματα, μία που έχει να κάνει με ποσοτική εστίαση και μία ποιοτική. Ποσοτικά. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Αλλά δεν λέει συγκεκριμένα πόσα δεν τολμάμε να πούμε κάποια, να θεσπίσουμε κάποια ποσοτικά κριτήρια για την απαραίτητη αύξηση του προϋπολογισμού για να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή τη φιλοδοξία και που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πραγματικό ποσοτικό επίπεδο μεταρρύθμισης. Νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, μπορούμε να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ποσοτική ε, προσέγγιση. Έχουμε το νομικό όριο, το 1,29% του ε, προϊόντος του ακαθάριστου προϊόντος Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρείται ότι είναι ανεδαφικό. Η Κομισιόν ποτέ δεν θέλησε να πλησιάσει αυτό το όριο βέβαια. Στην πρόταση της ε, στην πρόταση που έθεσε. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που έχουμε τώρα, είναι ουσιαστικά το κατώτατο όριο στο οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ο προπολογισμό και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη σε μια ποσοτική προσέγγιση. Ποιοτικότερα τώρα, σε ποιοτικό επίπεδο, πρέπει να προετοιμαστούμε για να υπάρξει μια πίεση από όλε τι ε, επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολιτισμός, ε, περιφερειακή, δεν πρέπει εμείς να αμυνθούμε εναντί αυτών των επιμέρους επιτροπών. Θα πρέπει να ενσωματώσουμε τις διεκδικήσεις τους που είναι απόλυτα θεμητές οι αιτήσεις τους. Πώς πρέπει να το κάνουμε τώρα αυτό. Η μεταρρύθμιση μας θα πρέπει να συγκλίνει και πάλι, να οδηγήσει και πάλι σε σύγκληση με την στρατηγική Ευρώπη 2020. Δεν πρέπει να την αφήσουμε μονάχα σε μια απότερη ρητορική αναφορά. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να την τηρήσει η πολιτική προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το ίδιο και το ελεκτικό συνέδριο στην έκθεσή του του 2014 είπε σαφώς σε ποιο βαθμό ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν επαρκώ συνεκτικός και συμβατός με τη στρατηγική 2020 Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό επίση μια άλλη παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ένα άλλο σημείο συγκεκριμενοποίησης, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενσωματώσουμε τις διεθνείς μας ε, υποχρεώσεις σε δύο τομείς, την COP21. Εδώ δεν υπάρχει μονάχα δεν υπάρχει θέμα συζήτηση, αλλά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις δεσμεύσει μα για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη για πάνω από 1,5% και επίσης θέλουμε να έχουμε μία λύση για τις ε, ε, μορφές ε, ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται ως ε, ε, εναλλακτική στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου. Και επίσης Χρειαζόμαστε και νέε προοπτικέ στον τομέα τη βιομηχανική πολιτική. Η Ευρώπη χρειάζεται μια αυθεντική βιομηχανική πολιτική που δεν έχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνει ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Είναι δυνατό να συζητήσουμε <coughs> αν θέλουμε να έχουμε ένα νέο ταμείο, μια μεταρρύθμιση των νομικών βάσεων, αν θέλουμε να κινηθούμε προς τις γραμμές της ε, ε, προσαρμογής ε, σε ενεργειακό τομέα, της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης κτλ. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά, αλλά δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει ο κύριος Κατάινον, ότι η πολιτική της ε, πολιτικής συνοχής να περιλαμβάνουν κριτήρια που έχουν να κάνουν με το Ταμείο Juncker, αλλά δεν έχουν να κάνουν με τον προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε την πολιτική συνοχή για να γίνει πιο συμβατή με τους στόχους του, της Ευρώπης 2020 και του COP21 και τέλος στοιχεία για την ε, μεταρρύθμιση μετά από το 2020. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσουν να, να μην ε, μιλήσουμε για το θέμα του ορίου των ε, ιδιών πόρων. Αυτό πρέπει να είναι στοιχείο της συζήτησης μετά το 2020. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ταμπού σε αυτή τη συζήτηση. Και δεύτερον, η μεταρρύθμιση των ιδιών πόρων βάσει της, ε, του πνεύματος των συνθήκων και αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα, να ζητήσουμε ότι η μορφή της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους δεν αποκλεί φόρο επί των εκπομπών άνθρακος ή φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή άλλες μορφές ε, φόρου για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Πρέπει τώρα να πούμε ότι το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι μία μορφή διευκολύνσεων σε φορολογικό επίπεδο, tax rulings, που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένα κράτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τις διατηρήσουμε αυτές τις διευκολύνσεις, αυτές τις απαλλαγές που παίρνουν ορισμένα κάτι μέρη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πεπαλαιωμένες αυτές οι ιδέες και έτσι αλλιώς οδηγούν σε μια ανισότητα και έλλειψη δικαιοσύνης του προϋπολογισμού. Κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε κύριος Ζάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές γιατί η έκθεσή τους είναι μια πολύ καλή βάση εκκίνησης για την πολύ σημαντική συζήτηση στην οποία πρέπει να αποδεθούμε. Εγώ συμμερίζομαι εν μέρει αυτό που είπαν οι προαναλύστοντες σε ό,τι αφορά τις βασικές υποθέσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν ήδη να δούμε πώς το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει περάσει μια πάρα πολύ ραγδαία εξέλιξη λόγω των γεγονότων, λόγω των πραγματικών συζητικών, λόγω των προκλήσεων που βλέπουμε κάθε μέρα. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα πρόβλημα, πάντα προσπαθεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια του προπολογισμού. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει, αυτό είναι ένα πρόβλημα για δύο λόγους. Για ένα πολιτικό λόγο, γιατί όλοι μας ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι σε μια κατάσταση πίεση των εθνικών προϋπολογισμών είναι να ζητήσουμε πρόσθετους πόρους για να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα και υπάρχει και ένα οικονομικό χρηματοπιστωτικό πρόβλημα στο, το οποίο μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν όταν μιλήσαμε με την κυρία Καλβίνιου. Δηλαδή έχουμε κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε αν χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων επιτρέπει την επιτεύξη των στόχων που θέλουμε ή θα ήταν καλύτερα να γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε και από τη βάση του εγγράφου αυτού, το οποίο αφορά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, θα πρέπει να είναι κατά πόσο ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρόσφορο εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση των μεταναστών, αν είναι το κατάλληλο εργαλείο για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας, αν είναι το σωστό εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου είναι μια ευκαιρία για να, είμαι, να είμαστε πραγματικά ρεαλιστές και να κρατήσουμε μπροστά από τα μάτια μας ένα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχουμε λοιπόν ένα προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το θέμα δεν είναι αν εμείς σαν Ευρωβουλευτές ζητάμε περισσότερα ή λιγότερα. Η δική μου αίτηση είναι ότι θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του κατά πόσο ένας πιο ευέλικτος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εφανερότητα με τις αυτές και τις αιτήσει που έχουμε κάθε μήνα, κάθε μήνα ή κάθε χρόνο, Έχουμε δυσκολία να ικανοποιήσουμε λοιπόν όλες αυτές τις αιτήσει. Πρέπει να βρούμε με έναν τρόπο λοιπόν να έχουμε καλύτερη ανταπόκριση στις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όπως ελέγχθη η διαπόρεση με τους ένα άλλο σημαντικό θέμα θα πρέπει να είναι η στέρηση στις πληρωμές που να συνδέεται πάντα με το θέμα των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Να κατανοήσουμε το να συνεχίσουμε με αυτό το χάσμα την υστέρηση μεταξύ πιστώσεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών σίγουρα δεν σταθεροποιεί, δεν επιλύει τα προβλήματα που έχουμε ενώπιον μας. Να μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι πολλές φορές ζητάμε πολύ περισσότερα από τον προπολογισμό από ό,τι μπορεί να αποδώσει. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει περιθώριο για ορθολογικοποίηση των πόρων που έχουμε αυτή τη στιγμή και είναι απαραίτητο να εστιάσουμε περισσότερο σε μερικούς εφικτούς και συγκεκριμένους στόχους ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πώ προσφέρει προσθέμενη αξία ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνω για ένα θέμα το οποίο για μένα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο τελικό κομμάτι τη συζήτηση όταν θεσπίσουμε τι βάσει για τον επόμενο πολιετή δημοσιονομικό προπολογισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση και σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή μας για μια μελλοντική δημοσιονομική εξουσία για την ε, Ευρωζώνη, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα έλθει στην επιφάνεια. Και ελπίζω ότι μαζί σας είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για τις προτάσει που θα διαμορφώσουν τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση. στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόλμια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολύ έπαινοι για τους δύο εισηγητές. Μου είναι δύσκολο, λοιπόν, να βρω νέο τρόπο να τους επενέσω, νέα λόγια. Είναι εντυπωσιακή η δουλειά που έχουν κάνει και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο με το σχέδιο κειμένου. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα. Καταρχάς, η έκθεση αυτή δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτα να επανεξετάσουμε τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο, στο δημοσιονομικό πλαίσιο και από εκεί να εξάγουμε συμπεράσματα για την αναθεώρησή του. έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι τα μέσα ευελιξίας μας έχουν εξαντληθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματισμός μας ε, μέχρι τώρα δεν ε, ήταν πολύ επιτυχημένος, δεν θα έπρεπε να έχουμε εξαντλήσει ήδη όλα τα μέσα ευελιξίας που είχαμε. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε προσεκτικά. Όταν έχουμε νέα καθήκοντα, νέα προγράμματα, χρειαζόμαστε είτε νέα κονδύλια είτε νέες προτεραιότητες. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να λειτουργήσει διότι αλλιώς ε, καταλήγουμε ακριβώς στο πρόβλημα των λογαριασμών που δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Και η επιλογή ανάμεσα στους ε, νέους πόρους ε, ή στις νέες προτεραιότητες όσον αφορά το δίλημα αυτό είναι η πιο ωραία απάντηση το να πούμε θα έχουμε νέα κονδύλια. Αλλά Κυρίε και κύριοι, αν δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι λάθος να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση, να σας ε, δώσω απλά ένα παράδειγμα. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το αν θα παραμείνει ή όχι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε στην Αυστρία ότι το FPÖ ε, ε, είχε ε, εκλογική νίκη. Βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι, ε, τα κόμματα που έχουν ε, σύνθημα λιγότερη Ευρωπαϊκή Ένωση ή καθόλου Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα έχουν επιτυχίες στις εκλογές. Δεν έχει λοιπόν νόημα να πούμε ότι όλα θα είναι εντάξει αν απλά έχουμε περισσότερους πόρους και απαιτήσουμε τα νέα αυτά κονδύλια από τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει είτε νέα χρέη είτε ε, περισσότερη φορολόγηση των ε, πολιτών. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα πάει στραβά. Δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, θα πρέπει ε, να επιμείνουμε σε αυτό για να είμαστε ρεαλιστές. Γι' αυτό όχι νέα έσοδα, όχι νέους ίδιους πόρους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τη διχάσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που βρίσκω πολύ καλά στην έκθεση αυτή. Για παράδειγμα ότι υπάρχει σκέψη για πενταετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και επίσης ότι θα πρέπει εγκαίρως να έχουμε διάλογο με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμένα μου αρέσει η έκθεση αυτή. Γιατί πέρα από το ότι απαριθμεί όλα τα πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζουμε και ε, ε, που αποτελούν πρόβλημα, ε, μας δείχνει ότι δεν ε, θα πρέπει να, υπολογίζουμε, να κάνουμε τους υπολογισμούς μας χωρίς ε, τον ε, ξενοδόχο. Θα πρέπει να σκεφτούμε τα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μία σύνοψη όλων όσων θα θέλαμε, αλλά δεν μας βοηθάει απλά να απαριθμούμε τις επιθυμίες μας. Αυτό που λείπει είναι το από πού μπορούν να προέλθουν τα χρήματα, από τα διαρθρωτικά ταμεία δηλαδή τα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή έχουν ε, τα μεγάλα μερίδια θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτα, διότι μόνο από εκεί μπορούμε να έχουμε τους σπόρους. Διότι αλλιώς έχουμε έναν ε, ατέρμονο ημάντα, θα πρέπει ε, να έχουμε συνεχή ανακατανομή των κονδυλίων. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από κάτι τέτοιο, από ένα τέτοιο φαύλο κύκλο για να αποφύγουμε και πολλές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Καλώς λέει ο Καλώς είπα, λέει ο πρόεδρος. Πολλοί έχουν θέσει ερωτήματα. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Και εγώ θέλω να χαιρετήσω αυτό το έργο, το ομαδικό, το οποίο είναι πολύ ρεαλιστικό και να τονίσω πώς είναι απαραίτητη πολιτική αναγκαιότητα η μεταρρύθμιση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αν δεν το κάνουμε θα, έρχο, θα έρθουν ακόμα λιγότεροι εκλογείς στις εκλογές του 2019. Θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι για την καθημερινή της ζωή. Γι' αυτό τον λόγο ορισμένοι θέλουν να φύγουν από την Ευρώπη γιατί δεν βλέπουν τελικά τι αντίκτυπο έχει η Ευρώπη στην καθημερινή της ζωή. <clears throat> αυτό οδηγεί στο Brexit, αυτό οδηγεί στην ε, ψήφο προς τα κόμματα ακραίων παρατάξεων και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επίπεδο πολιτικής. Οι πολίτες λοιπόν έχουν σαν να έχουν μπουχτίσει λιγάκι για την Ευρώπη. Σαν να είναι η Ευρώπη η οποία θα λύσει τα προβλήματα των ε, τα θέματα της ε, ευρωζωνικής ε, ε, ευρυζωνικού ίντερνετ. Μιλάμε συνέχεια για την ανεργία των νέων, μιλάμε συνέχεια για την ε, μικρομεσαίες και για τους νέους και όλα αυτά τελικά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε όλες αυτές τις αιτήσει των πολιτών. Θα πρέπει να είμαστε σοβαρή σε σχέση με τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι, ότι ε, υπογραμμίζονται οι βασικές αρχές, οι αρχές του, της οικουμενικότητας, της ενότητος της ενιαυσιμότητας, του προπολογισμού, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο αρχίζει να μας απασχολεί, ότι αυτός ο προπολογισμό ουσιαστικά δεν εξωτερικοποιείται. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια εξωτερήκευση η οποία εκφεύγει τελείως του δημοκρατικού ελέγχου. Για το θέμα των ιδιών πόρων ελέγχθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάποιο σημείο. Η Επιτροπή Μόντι μας είχε πει πολλά πράγματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, φοροδιαφυγές και φοροαποφυγές. Και ο κύριος ε, Μανκά αναφέρθηκε και στο θέμα του, της νομισματικής πολιτικής της ε, ρήψης από ελικοπτέρου, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, χρημάτων. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο προκαλεί και ορισμένα ε, ερωτήματα. Μήπως θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να έρθει εδώ ο κύριος Δράκη να μας πει ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμών ποια είναι η ιδέα του για την ελικοπτέρωση των χρημάτων. Εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε πάρα πολύ χώρο συζήτηση για τα θέματα αυτά, να είμαστε σοβαροί στα θέματα του προπολογισμού, αλλά ας δούμε και τα θέματα της νομισματικής πολιτικής που δεν είναι άμυρα σύνδεση με τα θέματα αυτά και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μάνκα ότι και εκεί υπάρχει μια δυνατότητα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Ωραία λέει ο πρόεδρος. με ένα καλό εκτυπωτή μπορούμε να δημιουργήσουμε ίδιους πόρους. Ναι. Ε, νομίζω ότι έχω εξαντλήσει τους εγγεγραμμένους ή όχι. Ζητήθηκε και από την Κομισιόν να εκφράσει την απόψή της, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι σχετικά. Αν θέλει να μας παρουσιάσει κάποια πρόταση. Μήπως μπορείτε να μας πείτε και πότε θα κάνετε κάτι τέτοιο. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο εξώμα της Κομισιόν. Κυρία Διευθυντά, παρακαλώ. με χωρίς μικρόφωνο μιλτής. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριοι Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε με ενδιαφέρον το σχέδιο έκθεσής σας. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή επανεξετάζει τα επιμέρους προγράμματα και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση ούτε για το πρόγραμμα, ούτε για το χρονοδιάγραμμα, συγγνώμη, ούτε για το περιεχόμενο της, ε, του αποτελέσματος της αναθεώρησης, ούτε όσον αφορά τις ε, σχετικές προτάσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Αντιπρόεδρο ε, έχει ραντεβού εδώ στην Επιτροπή σας για να συζητήσει την έκθεση όταν θα έχει σταθεροποιηθεί πολιτικά. Περιμένουμε προς το παρόν και θα σας ε, δώσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία όταν τα έχουμε και εμείς στη διάθεση. Ευχαριστούμε για αυτές τις ε, διευκρινήσεις. Μας καθυσυχάσατε. Μην, μην ε, το Παίρνετε άσχημα αυτό που λέω. Δεν δύναται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει να περιμένουμε, λέει, την 23η Ιουνίου. Οι συνάδελφοι Τωμά και Όλμπριχ πάντως παρόλα αυτά τα πέρασαν μια χαρά στην Επιτροπή μας σήμερα πιστεύω. Φιλοφρονήσεις έπεσαν βροχή και ήταν ομόφωνη η έπαινη των συναδέλφων προς τους δύο συνεισηγητές. Θα πρέπει το ευκταίο να γίνει και εφικτό είπε η κυρία Γκρέσλε. Όχι, όχι, τι είπε, ε, τι είναι δυνατό, τι είναι εφικτό. Αυτός ο στόχος της πολιτικής, να υλοποιείται το εφικτό. Εμεί θέλουμε να μάθουμε από εσά, μέσα ε, από του συνεισηγητέ, ε, από το ευθείο τι είναι εφικτό. Ε, κυρία Τωμά, ευχαριστώ, ευχαριστώ για, τις, ε, για τα ευγενή σα σχόλια και τι φιλοφρονήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους συναδέλφου για την υποστήριξή τους και να ευχαριστήσω τη γραμματέα, τη γραμματεία συγγνώμη, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και των πολιτικών ομάδων μας υποστήριξαν στη δουλειά μας και τους ευχαριστούμε. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση, είναι προφανές αυτό και καλό είναι να ε, τροφοδοτείτε και να διαρκέσει όσο χρειάζεται η συζήτηση και γι' αυτό διορθώστε με πρόεδρε. Ξεκινήσαμε ανάντητη δουλειά για αυτή την έκθεση περιμένοντας ε, στοιχεία από την Επιτροπή και καλά κάναμε από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, και για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν ξέρω, μήπω δεν ε, επιδέχεται και βελτίωσει το κείμενο, ε, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και βοηθήστε μας με τις τροπολογίες. Έλεγα λοιπόν ότι, ε, όπως ε, μας ρώτησε ο κύριος Φερνάντες, πρέ, ζήτησε και ο κύριος Φερνάντες, συγγνώμη, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το χρονοδιάγραμμα, ώστε αφενός να έχουμε το το την πενταετία αυτή περίοδο, αυτό το χρονοδιάγραμμα που επιτάσσει το, η εντολή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να, και να συμφιλιώσουμε αυτή την πενταετή περίοδο με τις ανάγκες του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου. Ε, και τον ε, ε, ΟΤΑ και γι' αυτό ε, ε, εισηγούμαστε εμείς αυτό το μεικτό σύστημα. Δηλαδή, αφενός έχουμε την πενταετή περίοδο, αλλά λέμε 5 συν 5 του τέστην 10 χρόνια με διάμεση αναθεώρηση. Έτσι, ανταποκρινόμαστε και σε αυτά που ζητάει η κυρία Μούτη ούτω ώστε όλε οι πολιτικέ, και δεν τι απαριθμούμε όλε, όλε οι πολιτικέ που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητε σε μακροπρόθεσμα να καλύπτονται. Και θα πρέπει ενδεχομένω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι μέσα στο κείμενο, όμω το μεικτό αυτό σύστημα κατά τη γνώμη μα καλύπτει τι ανάγκε. Δεύτερον, ε, δεν μπορώ να σχολιάσω όλα όσα είπε ο γιατί ε, ήταν πολλά. Ναι, όντω ε, μιλάμε για το 1β και όχι για το 1α. Για το 29 μιλάμε για το περιεχόμενο. Μετά την τροπολογία σας, ε, θα, αν καταθέσετε την τροπολογία, θα προσθέσουμε τα περί 2020, τον ορίζοντα 2020 και το ΣΕΦ. Τέλος πάντων, πέραν από ε, αυτών των σημείων θα ήθελα να σχολιάσω όλους ιδιαίτερα στο ζήτημα της ευελιξίας. Πολύ το αναφέρατε και όντω είναι πολύ συζητημένο το ζήτημα και όντω δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μία μεσοβέζικη λίγο στάση. Και γιατί το λέω αυτό, διότι και το διαπιστώσαμε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ε, ε, διότι λοιπόν ναι, μεν είναι απαραίτητη ευελιξία, όμως εγκυμονεί κινδύνους. Ε, όπως αυτόν που ανέφερε ο κύριος Φερνάντες, παραδείγματος χάρη, για το σχέδιο Γιούγκερ ήταν πολύ χρήσιμη η ευελιξία Φερρυπίν. Όμως ταυτόχρονα οδήγησε σε περικοπές προγραμμάτων, ε, κάτι που απευχόμαστε ουσιαστικά. Οπότε, επειδή σε ένα πλαίσιο Όντως χρειάζεται περιθώριο ευελιξίας, όντως χρειάζεται ένα περιθώριο ελιγμών, ε, το διαπιστώνουμε αυτό, αλλά για το τμήμα 3, 4 και 1β, κύριε Ντεπρέ, και κύριε Κιόλμεν, ναι, είναι ε, προτεραιότητες που αναγνωρίζονται από όλους όλοι αναγνωρίζουν ότι οι επενδύσεις, η καταπολέμηση ενεργείας των νέων, όλα αυτά συνιστούν προτεραιότητες. η ε, αναπτυξιακή βοήθεια, η βοήθεια προς τη, στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας, όλα αυτά θεωρούνται δεδομένα όμως. Αυτή η ευελιξία δεν σχετίζεται με μια μετεξελισσόμενη κατάσταση. Είναι σταθερέ οι ανάγκε μας, τουλάχιστον για τη διάρκεια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, και κύριε πρέπει να σας πω ότι ξυπακούεται ότι θα περιστρέφεται γύρω από αυτά τα ζητήματα η κατάσταση, ε, η συζήτηση, συγγνώμη, ε, αλλά ε, θα συζητήσουμε και το θέμα των χρηματοδοτικών μέσων και την ευελιξία που μπορούμε να έχουμε. Είναι προφανές. Αυτά μπορώ να σας απαντήσω προς το παρόν. Τώρα, για το πολιτικό θέμα, δηλαδή η χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων, ε, ε, πρέπει να εγγράφονται όλα αυτά μέσα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλέον ενδεδειγμένο μέσο ναι ή όχι. Όπως ε, λέω συχνά, είναι πολιτικές αποφάσεις. Κύριε Ολμπρίχτ, θέλω να μιλάω και για εσά, όμω θεωρώ ότι οι φιλοευρωπαίοι θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικότερο ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποδοχή των προσφύγων, ή για την προστασία των συνόρων, ή για την ασφάλεια, από ότι ένα εθνικό προπολογισμό. Και φυσικά οι αντιευρωπαϊστέ θεωρούν ότι για τα σύνορα καλό είναι να έχουμε ένα εθνικό προπολογισμό. Φυσικά, φυσικά θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Και παρότι δεν είστε ιδιαίτερα φιλοευρωπαίος, αναγνωρίστε παρακαλώ το ότι το ότι ε, μία ή δύο χώρες ε, είναι τα, τα πρώτα σημεία όπου έρχονται ε, οι πρόσφυγες για να μπουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες με το δικό τους προϋπολογισμό. Είναι οι πόρτε Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, κατά το ελάχιστο χρειάζεται Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για να συνδράμουμε αυτές τις χώρες που αντιμετωπίζουν αυτά τα προσφυγικά κύματα. Ε, Φυσικά, ανάλογα με τη στάση που έχουμε ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει κάποιο να παραμείνει εντό ή να βρεθεί εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλε απαντήσει θα δώσει στα προβλήματα που τίθενται και να πω ότι Συμφωνήσαμε με τον κύριο Όλμπριχτε να μην αναφερθούμε στο θέμα της Ευρωζώνης και των ε, δυνατοτήτων της, όχι μόνο διότι ε, ε, καταρτίζεται τώρα μια έκθεση που θα καλύψει αυτά τα ζητήματα, αλλά διότι το θέμα μας δεν ήταν αυτό. Το θέμα μας είναι η αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και ελπίζουμε να μην φύγουμε εκτός θέματος με τις τροπολογίες σας. Αυτό είναι το ε, βασικό μας σχέδιο, το Plan A που λέμε. Αν ε, αποτύχει αυτό και αν ε, το απαραίτητο δεν, συμπέσουν, δεν συμπέσει με το εφικτό, τότε θα προκύψει το εφεδρικό το σχέδιο με την Ευρωζώνη. Ευχαριστούμε κυρία Τωμά, λέει ο Πρόεδρος, για το θέμα του το προσφυγικό. Μην ξεχνάτε, στις 15 Ιουνίου έχουμε σημαντικότατη ακρόαση. Ε, οι συνάδελφοι από τη ΛΥΜΠΕ, από την ΑΦΕ θα έρθουν, είναι κοινή ακρόαση και νομίζω, κυρία Τομά, θα καλυφθούν οι ανάγκες που προαναφέρατε. Για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αύριο το πρωί σε έχουμε έχουμε μεικτή συνεδρίαση, ακριβώς για να δούμε ποιος θα μπορούσε να είναι ένας προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Όλμπριχτ. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω την πολωνική γλώσσα γιατί βλέπω όλους τους συναδέλφους μου να χρησιμοποιούν τις εθνικές τους γλώσσες. Ωραία, ωραία γλώσσα είναι και τα πολωνικά, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Σας ευχαριστώ. Komisja w tej, w tej sprawie, ponieważ uważamy, że Komisja Europejska czeka na wynik referendum brytyjskiego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 Νομίζω λοιπόν ότι το δημοψήφισμα στην ε, Ιταλία, θα μας, <clears throat> στη Μεγάλη Βρετανία, θα λύσει κάποια προβλήματα. Αλλά και εδώ και η Κομισιόν δεν θέλει να πάρει θέση, γιατί βλέπω ότι η Κομισιόν αναμένει τα αποτελέσματα του δημοψήφισματο για να σταθμίσει τη θέση τη. Δεύτερο θέμα. Θέλω να σα ευχαριστήσω για όλου του επένου. Θα ήταν καλό να έχουμε συμφωνία όλοι, όχι επειδή το ψήφισμα μας είναι τόσο ανούσιο και γενικό να το δέχονται όλοι, Ελπίζω ότι η επενή σα και η υποστήριξή σα δείχνει ότι έχουμε κάνει σωστά την εργασία μας μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν σημεία πολιτικής θέση που θα πρέπει να υπάρχουν στην ε, έκθεσή μα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόλμελ, με τον οποίο πάντα συζητώ για τα θέματα της προσέγγιση στο προπολογισμό. Είναι πολύ διαφορετική η θέση του κυρίου Κόλμελ με τη θέση του κυρίου Τσάνη αλλά είναι σαφείς προσεγγίσεις, διάφανες προσεγγίσεις και με τον τρόπο αυτό πρέπει να διακρεώσουμε το πολιτικό μας έργο για να υπάρχει σαφήνεια επί των θέσεών μας και με την βάση αυτή να λειτουργήσουμε. Τώρα, ο Γιάννος Λεβεντόφσκι έθεσε ένα σημαντικό θέμα. Γιατί να μην γίνει πρώτα η μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού πριν τελειώσει το πρώτο μισό της περίοδου προϋπολογισμού. μετά από το πρώτο εξάμεινο του 2017 θα πρέπει να γίνει η μεταρρύθμιση, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει η Κομισιόν να παρουσιάσει μια νέα πρόταση για το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε λοιπόν τώρα να υποχρεώσουμε την Κομισιόν να προετοιμάσει ένα έγγραφο μέχρι έχουμε την να προετοιμάσει η Κομισιόν το, την πρότασή της αυτή μέχρι το 2016. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά μόνο να περιμένουμε και αυτή την πρόταση. Αυτό που κάνουμε εμείς ως συζητητές καταδεικνύει ότι είναι απαραίτητο να γίνεται η μεταρρύθμιση πριν εκπνεύσει το πρώτο μισό της δημοσιονομικής ε, περίοδου. Πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό, αλλά σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουμε οριστικά αποτελέσματα, οριστικά πορίσματα και είμαστε υποχρεωμένοι από τη μορφή του προπολογισμού να αντλούμε τα συμπεράσματα ενώ είναι να εκτελέσει ο προπολογισμό. Επίση, ελέγχεται από πολλού ότι είναι απαραίτητη μια απλοποίηση. Και εδώ υπάρχουν νέε διατάξει οι οποίε αφορούν τι πολιτικέ μα. Εμεί έχουμε αποφασίσει να έχουμε μια σειρά από κατεξουσιοδότηση πράξεις. Κάποιες από αυτές έχουν μόλις δημοσιευτεί, άλλες δεν είναι ακόμα έτοιμες. Βρισκόμαστε στο τρίτο έτος λειτουργίας των δημοσιονομικών προοπτικών και οι αντίστοιχες ε, κατεξιότητες πράξεις έχουν δημοσιευτεί, έχουν εκδοθεί μόνο πριν από δύο τρεις Πώς θα λειτουργήσουν τα προγράμματα επιτοπίως αν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα απαραίτητα έγγραφα για να αρχίσουν να λειτουργούν τα προγράμματα. Ε, είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για απλοποίηση αν τελικά το αποτέλεσμα είναι να ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το δημοσιονομικό κανονισμό για να μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει να δούμε πού καθυστερήσαμε και πού είναι απαραίτητο να κάνουμε πιο γρήγορες τις διαδικασίες που είναι πραγματικά επαχθείς. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα ε, πιο γρήγορα και δεν θα πέσουμε στην πεγίδα που έχουμε στήσει τον εαυτό μας. Και τώρα για να απαντήσω στον κύριο Μαραγάλη ο οποίος ρώτησε γιατί δεν θέτουμε και αριθμητικά στοιχεία στην έκθεσή μας. Για μένα νομίζω ότι είναι η αρχή της συζήτησης, δεν είναι μια φάση στην οποία μπορούμε ήδη να αναφερθούμε σε αριθμητικά ποσά. Είναι η αρχή ενός διαλόγου και εξάλλου περιμένουμε και την πρόταση της Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν είναι αυτή η οποία έχει τα αριθμητικά στοιχεία, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται. Αν το κάνουμε λοιπόν πολύ πριν από το Δεκέμβριο, αυτό θα οδηγήσει ναι μεν στο να δείξουμε ότι είμαστε φιλόδοξοι, αλλά θα μας πούν ότι δεν ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αλλά για την COP21 επί τη, επί τη βάση των ε, πληροφοριών μας δεν υπάρχει εκτίμηση του κόστους για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Εάν είχαμε κάποια πληροφορία σχετικά θα την είχαμε συμπεριελάβει, αλλά βρίσκεται ακόμα στη φάση της κύρωσης της συμφωνίας. Δεν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα γι' αυτό. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε ακόμα να τα περιλάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία πλήρω. Ευχαριστώ κύριε Ολμπρίστε. Κλείνουμε την συζήτηση αυτή, η οποία ήταν εξαιρετικά πλούσια. Καταλάβαμε που είναι τα διακριτικά ε, πλαίσια για την Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει μέχρι τα τέλη Ιουνίου, εν η κυρία Τωμά και ο κύριος Ολμπριχτ και ο καθένας από εμάς με ήττα. Δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι δεν έχουμε ασκήσει την ασφικτική πίεση που χρειάζεται στην Κομισιόν, ώστε μέσα σε λογικά χρονικά όρια να καταθέσει προτάσεις της. Είναι σαφή τα πράγματα. Περνάμε τώρα στην κυρία Μακή για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της για το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση για την υπόθεση Μωρή Global. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ τη μητρική μου. Η Γαλλία λοιπόν ε, θέλει υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση ε, για την εταιρεία Mori Global SAS. Ε, έγιναν πολλές απολύσεις. Η αίτηση υποβλήθηκε πέρσι από την ε, Γαλλία τον Νοέμβριο. Πάνω από 2.000 δικαιούχοι προβλέπονται στην αίτηση αυτή και οι εργαζόμενοι, ε, οι δικαιούχοι βρίσκονται σε όλη την Γαλλία. 8,5 εκατομμύρια θα είναι το συνολικό ποσό που ζητείτε. Και 60 και κάτι χιλιάδες ε, ζητώνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ε, στην ε, Παγκοσμιοποίηση. Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την ε, εξέβρεση θέσεων ε, εργασίας για τους ανθρώπους αυτούς. Το 2013 η Γαλλία πάλι είχε ζητήσει κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής ε, στην παγκοσμιοποίηση. Περίπου 4.000 άνθρωποι από την ε, επιχείρηση Mori Global ε, αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Η επιχείρηση προσπαθεί να βρει θέση εργασίας για 2.132 εργαζομένους και ακριβώς ε, για αυτούς ζητείται η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στη Παγκοσμιοποίηση. Η εταιρεία αυτή επηρεάστηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Η εισαγωγή προϊόντων μειώθηκε σημαντικά. Έχουμε περίπου 30% αύξηση των φορτηγών στις οδικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να έχει δραστηριοποιηθεί πιο γρήγορα, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων. Η επιχείρηση αυτή ουσιαστικά ζητά χρηματοδότηση ε, των ιδίων υπηρεσιών που χρηματοδοτήθηκαν ε, σε προηγούμενες περιπτώσεις κινητοποίησης ε, του Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι πληρούνται όλε οι, προ... προϋποθέσεις ε, για την κινητοποίηση του Ταμείου στην αίτηση αυτή. Ε, το Κοινοβούλιο μπορεί να υποστηρίξει την αίτηση αυτή. Ε, περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας και προθεσμία είναι τον Μάιο. Νομίζω όμω ότι κύριε Πρόεδρε εσείς γνωρίζετε καλύτερα την περίπτωση αυτή από ότι εγώ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε όλοι τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο τομέα των μεταφορών η Ευρώπη των μεταφορών, η ενιαία Ευρώπη των μεταφορών φυσικά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Οι εθνικές νομοθεσίες είναι διαφορετικές από τη μια χώρα στην άλλη και βλέπουμε φαινόμενα μετακίνηση επιχειρήσεων. Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θέτουν τις έδρες τους στις νέες χώρες, στη Βουλγαρία, Λιθουανία, Ρουμανία Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποιες είναι οι αντιδράσεις των συνάδελφων. Κύριε Μπένανο. Βεβαίω κύριε Πρόεδρε, είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω πολύ καλά. Γιατί και εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό της Μωρή Global. Μετά από τη Μωρή Δικρό δημιουργήθηκε η Μωρή Global. Δεν πέρασε όπως να καλύψει την ε, επιβίωσή της, γιατί όλος το τομέα μεταφορών είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και αυτό που είπατε κι εσείς. Υπάρχει η κοινωνική νομοθεσία σε κάθε χώρα που οδηγεί σε μια μορφή ανταγωνισμού προς τα κάτω, η οποία εμποδίζει τουλάχιστον τους Γάλλους μεταφορείς να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασκούν το έργο τους. Έχουμε τονίσει την ανάγκη να υπάρχει ο θεμητός ανταγωνισμός. Και μου λέγει ένας Ούγγρος συνομιλητής μου ότι τι θεμητός ανταγωνισμός όταν στην Ουγγαρία ο Ούγγρος γεωργός παίρνει τέσσερις φορές λιγότερο από το Γάλλο για τα ίδια προϊόντα, Πού βρίσκεται ο θεμητό ανταγωνισμό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξακολουθήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα αυτό, αλλά δεν προχώρησε και πάρα πολύ πρέπει να πιέσουμε για να μπορέσει να γίνει κάτι από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να εξακολουθήσουν να εργάζονται για αυτή την απαραίτητη εναρμόνιση, γιατί η μορή Global είναι θύμα του, της παγκοσμιοποίησης, όπως υπονοεί και το όνομά τη. Είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει δημοσιονομική, δεν υπάρχει φορολογική, αλλά και εργασιακή εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση αυτές, όπου ξέρουμε ήδη τι θα γίνει. Θα ήταν χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις να εργαστούν για περισσότερη καινοτομία και για να μπορούν να προλαβαίνουν τις εξελίξεις. Αυτό θα και εγώ να κάνω όταν παρουσιάσω την εκθεσή μου για τις μικρομεσαίες. Νομίζω ότι δεν αρκεί να καταλήγουμε σε μια διάγνωση και είναι σαφής η διάγνωση για την μόρη global αλλά είναι απαραίτητο να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι διεθνεί εξέλιξει, οι οποίε δεν επιτρέπουν να παράγουμε τα προϊόντα όπω πριν από 50 χρόνια και θα πρέπει να επιτρέψουμε στι επιχείρησει να κινηθούν προ άλλη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να σχολιάσει εδώ. Εγώ θα πω κάτι ο ίδιο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών. Εδώ μιλάμε για έσω-ευρωπαϊκή ε, προσαρμογή και όχι προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Ίσως εδώ θα έπρεπε να έχουμε και μια σημασιολογικού χαρακτήρα τροπολογία. Γιατί τα θέματα των μεταφορών, των οδικών μεταφορών είναι έσω-ευρωπαϊκά θέματα και είναι μια προσαρμογή στην ευρωπαϊκότητα και όχι στην παγκοσμιότητα. Του του λεχθέντος όμως θα ζητήσω από τον εισηγητή μας να κλείσει την, ε, <clears throat> τη συζήτηση για το, την εισηγητρία μας να κλείσει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Όλα ελέγχθησαν. Όλα είναι λελεχθέντα. Θα κατατεθούν οι τροπολογίες μέχρι τις 10 Μαΐου στις 12 η ώρα που είναι η καταληκτική προθεσμία. 23 Μαΐου στην Επιτροπή Προεπολευσμών θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό και θα ψηφίσουμε και στις 25 Μαΐου θα έρθει στην Ολομέλεια. Στρέφομαι προς την κυρία Χολμάιερ. Θέλετε να κάνουμε την ψηφοφορία αυτή που είχατε ζητήσει, κυρία Χολμάιερ, από ό,τι είχα καταλάβει. Θέλετε να υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία για το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, είχα μοναχα τρεις μέρες στη διάθεσή μου για να μπορέσω να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα θέματα, κάμια διακοσάρια σελίδες και μόνο. Μπορώ να σας πω σαφώς ναι, θα ζητήσω μέχρι τις 23 Μαΐου προθεσμία για να μπορέσω να εξετάσω καλύτερα τους φακέλους αυτούς γιατί υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες ελείπουν και για τα δύο κτίρια στη Μερότ και το Black Pearl νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια πρόσθετα στοιχεία και υπάρχει και ένα τρίτο κτίριο το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη και δεν ξέρω τώρα, δεν, δεν έχω κάποια στοιχεία γιατί το κτίριο αυτό, το τρίτο δεν περιλαμβάνεται. Υπάρχει ένα περιο, περιθώριο 8% για την ε, για τη Σύμβαση Χρησικτησίας, το οποίο μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ υψηλό. Γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω, επειδή μόνο τρεις μέρες είχα στη διάθεσή μου να διαβάσω τα κείμενα αυτά, να μπορέσω να θέσω κάποια ερωτήματα προς την Κομισιόν, γιατί και οι συνάδελφοι, ο Ζεραντέπρα και, ο, αυτός έχει ζητήσει να υπάρχει περισσότερος χρόνος, γι' αυτό θέλω να έχω την δυνατότητα να μπορέσουμε να <clears throat> έχουμε περισσότερα στοιχεία. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να έχουμε την ε, παράταση αυτή των δύο εβδομάδων. Για το δεύτερο θέμα έχουμε κάπως περισσότερο χρόνο. Είναι ένα τρίτο κτίριο για το Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Καλς Ρούι. το οποίο βρίσκεται σε μια διαδικασία που εμπλέκει τα θέματα της ε, ασφάλειας για την ε, πυρηνική έρευνα. 80% της έρευνας πραγματικά λαμβάνει χώρα σε αυτό το κτίριο και γι' αυτό τα εργαστήρια εκεί τα οποία είναι πεπαλαιωμένα θα πρέπει να επαναρρυθμιστούν για να μπορεί να γίνει πάλι σωστά <clears throat> η έρευνα αυτή. Αυτό σημαίνει ότι θα εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια από σεισμούς, από βόμβες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει η αναδιαμόρφωση των κτηρίων αυτών. Αυτό δεν έχει κάποια συνέπεια σε επίπεδο προϋπολογισμού γιατί έχουν το δικό τους προϋπολογισμό τα, τα κοινά κέντρα ερευνών και παίρνουν χρήματα και από τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν εκεί. <clears throat> Μπορούμε λοιπόν στις 23 Μαΐου και το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε γιατί έτσι θα έχω πραγματικά τη δυνατότητα να εξετάσω το κείμενο αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει πίεση για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε νωρίτερα και έχουμε πει για τα κοινά κέντρα ερευνών ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα ποσά για, τα, για τις απρόπτες περιστάσεις και νομίζω αυτή τη στιγμή έχουν γίνει οι, τελευταί, οι τελευταίες εργασίες που έγιναν στον τομέα αυτό έγιναν χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού, οπότε έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα γίνει το ίδιο και τώρα. Σας ευχαριστώ, λέει ο, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε, κυρία Χολμάιερ. Για την δουλειά που κάνετε, κατέχετε το θέμα σε κάθε λεπτομέρεια ε, για τα κτίρια, κυρίως Black Pearl και με Ε, νομίζω θα σε υποστηρίξουν για την 15η ε, ημερή παράταση, διότι όλοι θέλουν να γνωρίζουν το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και για να ε, τηρούμε ε, μια ε, σωστή νομοπαρασκευαστική διαδικασία νομίζω ότι καλό θα ήταν να χορηγηθεί αυτή η παράταση. Έχει πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ήθελα μόνο να πω πως για αυτά τα δύο κτίρια προβλέπεται στις 15 Μαΐου να υπογραφεί η σύμβαση. Σε 11 Απριλίου είχαμε τη γαλλική εκδοχή. Στις 24 Μαΐου 23 είναι η επόμενη συνεδρίαση της Κόμπου, οπότε ε, θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Ζητώ από την εισηγήτρια να ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Θα ε, βάλουμε τα δυνατά μας. Ε, κυρία Χολμαϊέ. Πολύ ευγενικά να πω στην Κομισιόν ε, πώς θα ήταν εάν εγκαίρως κάνατε τις παρουσιάσεις ώστε να τις προλαβαίνανε οι συγητέ. Η Κομισιόν ευθύνεται για την καθυστέρηση και οι συνάδελφοι δεν είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, υποβάλει τα πράγματα εγκαίρως, ε, διότι ακόμα και το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε μας το έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας είπε βρείτε εσείς τις απαντήσεις σας από 150 σελίδες. Νομίζω ότι δεν ήταν αρκετά η οι απαντήσεις σας. Ε, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν καθυστερήσαμε εμεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρησε. Επίσης θα ήθελα ε, να έχουμε παράταση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, μετά στον Όσων, το ECDC. Διότι έχουμε δύο εβδομάδες όπου δεν κάνουμε τίποτα, αλλά μην θεωρήσετε ότι ε, έχει εγκριθεί το θέμα αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν και στο σημείο αυτό δύο εβδομάδες, δύο εβδομάδες παράταση. Donc, euh, <laughs> plus, on m'a dit que pour CDC... Δεν ξέρω, να πω για το SNDC. Μόλις πήραμε το τρίτο σχέδιο αυτό. Έχουμε και μια ευθύνη που επομιζόμαστε. <clears throat> Θέλουμε να βοηθήσουμε την Κομισιόν, αλλά υπάρχει και ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά το έργο μας. Κύριε Πεζάνο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αν βρούμε την ευκαιρία, ίσως μέσα στις επόμενες 15 μέρες, αν μπορέσουμε να συνεδριάσουμε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δυνατό για να σεβαστούμε την ημερομηνία της 15ης Μαΐου Ασφαλιτός χρειαζόμαστε δύο εβδομάδες πρόσθετες. Και έχουμε ούτως ή άλλως την ε, παράταση κατά 19, μέχρι 19 Μαΐου. Αλλά είναι, εάν η Κομισιόν μας είχε δώσει το έγγραφό της νωρίτερα, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι απαραίτητο λοιπόν και δεν πρέπει η Κομισιόν να θεωρεί ότι εμείς φταίμε για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε το έγγραφο αυτό. Η Κομισιόν λοιπόν κάνει κάτι το οποίο πολλές φορές που μας θέτει σε πίεση χρόνου και μας υποχρεώνει να αναβάλουμε την, ε, ε, την ε, εξέτασή μας. Λοιπόν, αυτό δεν με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει να μας δίνουν γέρο στα έγγραφα. και πιστεύω νομίζω ότι αν δεν το ζητούσατε εσείς 19 Μαΐου συν δύο εβδομάδες, κάποιος από την Επιτροπή μας θα το ζητούσε. Αλλά ευτυχώς έχετε αυτή την πεποίθηση και το θάρρος γιατί ε, αν είχαν δοθεί εγκαίρω όλα αυτά τα έγγραφα, μπορούσαμε να ψηφίσουμε σήμερα. Θα πρέπει περιμένουμε λοιπόν, κυρία Χόλμα να κάνει την απαραίτητη ανάλυση <clears throat> και θα περιμένουμε μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή και για την επόμενη φορά, λοιπόν, κύριε Πρεζόνς. Αν μπορούμε να έχουμε λίγο ταχύτερα τα έγγραφα, αυτό θα είναι ένδειξη ευδιοίκησης, ευδιαχείρισης. Έχει τελειώσει λοιπόν η μέρα για διαταξή μας για σήμερα το απόγευμα. Αν δεν έχετε κάποιο άλλο θέμα, διακόπτουμε. Αύριο το πρωί στις 9 η ώρα σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων για το σχέδιο προϋπολογισμού της Ζώνης Ευρώ και εμείς εδώ στις 10.30 σε αυτή την αίθουσα θα είμαστε. Η κοινή μας συνεδρίαση με την ΕΚΟΝ θα είναι στο, έγραφο, στο ε, ε, κτίριο PPHS 3C50. Διακοπή της συνεδρίας μέχρι αύριο. Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι. Bon. Parfait. Donc demain, il y a des votes. Oui. Des débats